Καλημέρα. Να εγκρίνουμε πρώτα την ερήσια διάταξη. Υπάρχει κάποια παρατήρηση. Εγκρίνεται. Οπότε... Συνεχίζουμε με τα σημεία 2 έως 4 στην ημερήσια διάταξη που όπως ξέρετε αφορούν την εκλογή δεύτερου, τρίτου και τέταρτου αντιπρόεδρου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε τώρα σε θέση να προχωρήσουμε για να συσταθεί το Προεδρείο μας και να αρχίσει να λειτουργεί για ε, να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν χρειάζεται να σας πω γιατί αναστήλαμε την ε, εκλογή του Προεδρείου γιατί ένας κανόνας δεν είχε ευθυγραμμιστεί πλήρως ε, στην συμφωνία των πολιτικών ομάδων οπότε δεν ήμασταν σε θέση να εκλέξουμε Προεδρείο σύμφωνα με το άρθρο 204 παραγραφός 1 Νομίζω όμως ότι τώρα συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, να ονομάσω επίσης, να πω ποιοι είναι οι αναπληρωτές. Δεν με έχουν ενημερώσει από το ΕΛΚΑ, από τους σοσιαλδημοκράτες η κυρία Καηλή, η Βοτζάνη αντικαθιστή των Πολιτάν, Τσιμώνα Μποναφέ αντικαθιστά των Λουίτσι Μόργανο, Star Σταρμπάτη αντικαθιστά τον Μπέρντ Λούκε για το Άλντε Viernica αντικαθιστά την ε, κυρία Φανιβιον Δεν ε, βλέπω κάποιους άλλου να αναπληρώνουν, δεν με έχουν ενημερώσει. Τώρα. Δεν μπορούμε. Ε, έχουμε. Έχουμε απαρτία. Ε, ναι. Ναι, παρακαλώ. Έχω μπερδευτεί λίγο, δεν έχω πρόβλημα επί της ουσίας, απλά για να μην υπάρξει κάποια νομική αμφισβήτηση. Εγώ όπως αντιλαμβάνομαι τον κανονισμό, ε, οι αναπληρωτές πρέπει να είναι αναπληρωτές της ΕΚΟΝ ή μπορεί να είναι οποιοδήποτε βουλευτής. Δεν θέλω μετά να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα, έτσι θα ήταν πλακώδες. Όπως ξέρετε, υπάρχει η δυνατότητα για τις ε, ψηφοφορίες και άρα κατά αναλογία ε, και για τις ε, εκλογές ότι υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης από βουλευτή. Επί τη ευκαιρία όλοι μέλη της ΕΚΟΝ είναι που βλέπω εδώ, οπότε δεν υπάρχει το ζήτημα που αναφέρεται. Αλλά και να υπήρχε δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά τουλάχιστον τα ονόματα που διάβασα εγώ είναι όλοι αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Οπότε μπορεί να γίνει κάποια άλλη στιγμή αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, απαρτία έχουμε. Τώρα, υποψηφιότητες για την θέση του δεύτερου αντιπρόεδρου. Έχουμε κάποιες προτάσεις. Πέρβανς Μπερές. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προτείνω τον Πίτερ Σίμον. Uh, ναι, ευχαριστώ. Συμφωνεί ο υποψήφιος. Ναι. Το σημειώνω. Είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής. Έχει συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Προτείνω λοιπόν να εκλεγεί διαβοή. Συγχαρητήρια. Ελάτε στο Προεδρείο λοιπόν. Now we proceed... Uh, Περνάμε τώρα στην εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου. Υπάρχουν προτάσεις. Παρακαλώ. Και η Σουίνμπορν θα ήθελα να προτείνω. Σας ευχαριστώ. Η υποψήφια συμφωνεί. Επίσης είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής και έχει συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Νομίζω μπορεί να εκλεγεί διαβοής. Ευχαριστούμε, και Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Λοιπόν, ελάτε κι εσείς ανεβείτε στο βήμα. Και τώρα ζητάω υποψηφιότητε για την εκλογή του του πρόεδρου Μπουρκχαρτ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω τον συνάδελφο Λούντε Κνίτερμα εν του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ο υποψήφιο συμφωνεί. Είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής και έχει συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Συγχαρητήρια λοιπόν. Ωραίοτατα. Τώρα με πλήρες προεδρείο. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5, ανακοινώσει του Πρόεδρου. Να σα ενημερώσω για τους ε, τριμερεί διαλόγου. Ο τρίτος ε, για τα θέματα τη τυπλοποίηση έγινε την 3η 7 Μαρτίου. Σημειώθηκε σημαντική πρόοδο για το ΣΥΡΑΡ 5 Ζητήματα που αφορούν ε, το όριο των συναλλαγών σε επίπεδο προγράμματο. υπολογισμός τη αξία και έκθεση σε τιτλοποίηση, όμως ε, θα χρειαστούν περισσότερες συζητήσεις πριν συμφωνούσουμε για τις ενδιάμεσες ε, θέσεις ε, και τον, τη μεταφορά του κινδύνου. Για το STS πάλι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις απαιτήσει του προγράμματος για το πλαίσιο STS, αλλά οι συνομοθέτες είχαν διαφορετικές απόψεις για την διαδικασία πιστοποίησης το ρόλο των τρίτων μερών ιδιαίτερα και την εποπτεία της, ε, των απλών ε, αυτών τιτλοποιήσεων. Μετά από έκθεση των επιχειρημάτων συμφωνήσαμε σε μία μέθοδο να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε ένα πακέτο μέτρων ε, για να υπάρξει σταθερότητα στην αγορά τηλεοποίησης. Για την διαφάνεια πλησίασαν οι απόψεις μας, καθώς και οι δύο κλείναμε προς ε, τα αποθετήρια δεδομένων τιτλοποίησης, αλλά οι περαιτέρω λεπτομέρειες ε, για το ρυθμιστικό πλαίσιο και το ποιες πληροφορίες θα πηγαίνουν σε αυτά τα αποθετήρια ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε, αλλά θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την επικοδομητική συνεισφορά. Τέλος, το πολιτικό επίπεδο ενέκρινε την τεχνική εργασία και στους δύο φακέλους. Διάλογος έφερα 27 Φεβρουαρίου για τη συγχρηματοδότηση της ΕΦΡΑ και συμφωνήσαμε. Πολλές τροπολογίες του Κοινοβουλίου έγιναν δεκτές αυτές οι οποίες επιβάλλουν μεταξύ άλλων επιπρόσθετες υποχρεώσεις αναφορά στην Κομισιόν για το Ίδρυμα ΑΕΦΡΕΣ και την ΕΦΡΑΚ. Σας ευχαριστούμε κύριε Στόλικεν και ε, αναμένεται να συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή στην, ε, στις 22 Μαρτίου. Περνάμε τώρα στο σημείο 6 ισοδυναμία τρίτων χωρών, ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Καλώς ορίζω τον Όλιβιε Γκερσάν, τον Γενικό Διευθυντή της Τιτζεφίσμα και τους τρεις Προέδρους των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. I think it is a very timely and important... Πολύ επίκαιρη νομίζω η συζήτηση για ένα θέμα το οποίο βεβαίως είναι από μόνο του πολύ σημαντικό και προφανώς είναι στο κέντρο της ε, προσοχής ε, των διαπραγματεύσεων για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Περίπλοκο ζήτημα και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με τους συνομιλητές αυτούς. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι η Κομισιόν ε, υιοθέτησε μια ανακοίνωση προσφάτως. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με τον κύριο Κερσάν. Να σας δώσω τον λόγο για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Αγαπητοί ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε <clears throat> για να συζητήσω τη δουλειά που κάνει η Κομισιόν για το ρυθμιστικό καθεστώς των τρίτων χωρών. Είναι μια πολύ επίκαιρη συζήτηση. Στις 27 Φεβρουαρίου δημοσιεύσαμε ένα έγγραφο της Κομισιόν και έγινε μια καλή συζήτηση πρώτη με τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκι την περασμένη εβδομάδα επί του θέματος αυτού είναι αυτή η ισοδυναμία. Τα καθεστώτα τρίτων χωρών ήταν πάντα ένα σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίες και η προσέγγιση έχει εξελιχθεί ε, από όλη την νομοθεσία που, εγκρίναμε από τη χρηματοπιστωτική κρίση και μετά, πάντα διερωτηθήκαμε εάν είναι αρκετέ οι διατάξει ε, περί τη χώρα. Και οποτεδήποτε η απάντηση ήταν θετική, συνεργαστήκαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο για να αναπτύξουμε κατάλληλου κανόνε για αυτή την νομοθεσία ή για αυτά τα νομοθετήματα. Οι χρηματαγορές δεν είναι απλώ αγορέ, είναι παγκόσμιε αγορέ και δεν είναι προφανώς αγορέ μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως είναι πολύ σωστό να εξετάσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τους ε, ξένους φορείς και, η δράση που, έγινε ε, στο G20 με τα πρότυπα έγινε με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όποτε εφαρμόζονται οι διατάξεις τρίτης χώρας, ε, θα πρέπει να δούμε αν εφαρμόζονται ε, αποτελεσματικά τα διεθνή πρότυπα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό εξετάζουμε. Η ισοδυναμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέτει κάποιους προνοιακούς ε, προληπτικούς στόχους. Θέλουμε να αποφύγουμε τους περιττούς κινδύνους ε, και να τους εισάγουμε στο δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και όταν δεχόμαστε να τους εισάγουμε, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι ξένες δικαιοδοσίες τους διαχειρίζονται σωστά. Θέλουμε να αποφύγουμε το ρυθμιστικό αρμπιτράζ ή την παράκαμψη των κανόνων. Όποιο δεν παίζει με του κανόνε μπορεί μέσω των διασυνοριακών δραστηριοτήτων να δημιουργήσει πρόσθετου κινδύνου στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ορισμένε περιπτώσει, η ισοδυναμία μπορεί να μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε του περιτού και επιζήμιου ε, εξοεδαφικού αυτού παράγοντε λόγω των ξένων κανόνων ε, και η ισοδυναμία βασίζεται σε μια αξιολόγηση του ρυθμιστικού ε, και εποπτικού συστήματος των τρίτων χωρών. Ε, λαμβάνεται υπόψη εάν οι κανόνες αυτών των τρίτων χωρών επιτυγχάνουν τα ίδια ρυθμιστικά ή εποπτικά αποτελέσματα όπως οι δικοί μας κανόνες. Εάν δοθεί ισοδυναμία, τότε μπορούμε να εμπιστευτούμε τους κανόνες και την εποπτεία μιας ξένης δικαιοδοσίας σε ένα συγκεκριμένο τομέα ε, και να θεωρήσουμε ότι δεν δημιουργούνται κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την, τον τρόπο που κινούνται οι αγορές ή να δημιουργηθούν άλλοι κίνδυνοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά, ε, τα καθεστώτα ισοδυναμίας τρίτων χωρών έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τους σκοπούς ε, των κανόνων, τις παραμέτρους ε, που λαμβάνουν υπόψη για την αξιολόγηση ισοδυναμίας, τις, ε, την τεχνική συνδρομή των εποπτικών αρχών κτλ. Η προσέγγιση όμως που, που έχουμε είναι ότι λαμβάνουμε υπόψη του συγκεκριμένου αριθμιστικού στόχου του κάθε νομοθετήματο. Δηλαδή δεν έχουμε μία νομοθεσία, ένα νομοθέτημα που αφορά τι εξωτερικέ πτυχέ τη ενιαία ευρωπαϊκή αγορά στι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Ασχολούμαστε δηλαδή με την ισοδυναμία περιπτωσιολογικά. Φυσικά υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, ακόμα και μέσα στην Επιτροπή σα. Το έγγραφο εργασία ε, τη ε, Κομισιόν δείχνει ότι υπάρχει αυτό ο βαθμό ευελιξία και ότι έχει βοηθήσει τα καθεστώτα ισοδυναμία και έχουν αποδείξει αυτά ότι αξίζει να χρησιμοποιούνται. Ε, υπάρχουν δύο δέσμε προποθέσεων. Ε, ε Καταρχά, ελέγχουμε το πόσο είναι. Καταρχάς, ας πούμε, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το καθεστώ ε, εκθέσεων αναχώρα, τη πούμε, βιομηχανία. ε, έχει τελείω διαφορετικέ ανάγκες από τις, ε, τα στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψη μα για να δώσουμε ισοδυναμία ας πούμε, στους οργανισμούς ε, αξιολόγηση Πριν από δύο χρόνια ο προκατοχό μου έκανε μια αντίστοιχη συζήτηση με τα μέλη τη Επιτροπής σα. Ε, μίλησε για τη σημασία της αναλογικότητα ε, υπάρχουν δικαιοδοσίε που μα επηρεάζουν πάρα πολύ και άλλε ε, λιγότερο. Ε, αυτές που μας επηρεάσουν ε, λίγο ε, έχουν μικρή διεπαφή, μικρή ε, αλληλεπίδραση με τις δικές μας αγορές και αφήνουν ένα μικρό παγκόσμιο αποτύπωμα. Ενώ οι άλλες προφανώς μας επηρεάσουν περισσότερο. Όταν κάναμε, έγιναν αυτές οι παρατηρήσεις από τον προκάτοχό μου τότε, κάναμε συζητήσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες και θυμάμαι πολύ καλά ότι ο Στίβεν και εγώ είχαμε διάφορες δύσκολες συζητήσεις ε, για τις πρακτικές ε, εποπτείας των Αμερικανών, ας πούμε. Από τις αρχικές δημόσιες αντιδράσεις στο έγγραφό μας, από ό,τι φαίνεται η αναλογικότητα, φαίνεται, μοιάζει η αναλογικότητα να είναι ένα νέο χαρακτηριστικό. Αλλά όπως σας εξήγησα, υπάρχει. Πάντα είχαμε μια τέτοια προσέγγιση ε, σε ό,τι αφορά την ε, χορήγηση ισοδυναμίας στα καθεστώτα τρίτων χωρών. Και το έχουμε εφαρμόσει σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως στην περίπτωση με του Αμερικάνου που μόλι ανέφερα. Να σας εξηγήσω τι προσπαθούμε να πετύχουμε μέσω του εγγράφου αυτού. Στην πραγματικότητα είναι μια επισκόπηση με βάση τα στοιχεία που έχουμε, ε, της διαδικασίας ισοδυναμίας ε, με τρίτες χώρες ε, στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Είναι ένας απολογισμός που δείχνει πώς ε, η ισοδυναμία ε, λειτουργεί και προστατεύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ακαιρεότητα των αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διευκολύνει ε, την περαιτέρω ανάπτυξη των ολοκληρωμένων ε, χρηματαγορών. Είχαμε πάνω από 200 αποφάσεις για το θέμα αυτό και αποφασίσαμε να είμαστε πιο διαφανείς. Η έκθεση αυτή τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, να γίνει πιο αποτελεσματικό το πλαίσιο ισοδυναμίας. Ε, θα πρέπει ε, και να εφαρμόσουμε την αναλογικότητα και μια προσέγγιση που να βασίζεται στον κίνδυνο ε, και με βάση όλα αυτά να αξιολογούμε την ισοδυναμία. Θα πρέπει ο ρόλος των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών να ξεκαθαριστεί αξιολογώντας ε, το πλαίσιο, το ρυθμιστικό και εποπτικό των ξένων δικαιοδοσιών και να ξεκαθαριστεί η συμμετοχή στην παρακολούθηση και στην εφαρμογή ε, των αποφάσεων. Αυτή τη στιγμή δοθεί ε, θετική απόφαση ισοδυναμίας από την Κομισιόν. Δεν παρουσιάζουμε δηλαδή νέε προτάσει με αυτό το έγγραφο σε αυτή τη φάση. Ε, προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Κομισιόν σε διαδικασίε χορήγηση ισοδυναμία. Ε, Επίσης, οι συμμετέχοντες στην αγορά ε, πολλές φορές δεν καταλάβαιναν την ε, έννοια της αναλογικότητας και την ε, προσέγγιση μας βάσει του κινδύνου. Προσπαθούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε μια διαφάνεια. Επίσης, Πρόεδρε, πριν κλείσω, θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα του χρονισμού. Αναλύουμε καθεστώτα ισοδυναμίας εδώ και καιρό. Η πρόθεσή μας αρχικά ήταν να δημοσιεύσουμε αυτή την έκθεση πέρυσι πέρυσι στα πλαίσια μιας ε, μεγάλης προσπάθειας απολογισμού και καταγραφής της κατάστασης ε, στην νομοθεσία για τις χρηματαγορές. Όμως τελικά αναλύοντας τα καθεστώτα τρίτων χωρών χρειαστήκαμε πολύ περισσότερο χρόνο ε, για να λάβουμε υπόψη μας την αποτελεσματικότητά τους. Θα κάνουμε διάφοροι, θα συνεχίσουμε τη δουλειά φέτος επίσης θα ξαναδούμε κάποιες ε, προσεγγίσεις ε, για την ισοδυναμία τριτών χωρών με βάση την εμπειρία μας. Και όλα αυτά ε, τα κάναμε ε, στα πλαίσια της δουλειά που κάνουμε υπό την ηγεσία του Λόρδου Χιλ. Και φυσικά ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο περιμένουμε και τις ερωτήσεις σας και τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, Ολιβία Γκερσάν. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή. Στην επόμενη μιλήτρια μάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε. Όχι, στον επόμενο μιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αναφερθήκαμε λοιπόν σε αυτό το θέμα το οποίο είναι η προσέγγιση του θέματος της, ισοδυναμίας ε, για ε, σε τρίτες ε, χώρες ε, και βεβαίως αυτό βασίζεται στην, όχι ακριβώς στην μεταφορά του νομοθετικού πλαισίου σε κάποια άλλη τρίτη χώρα αλλά στη δυνατότητα στενής σύγκρισης ανάμεσα στις βασικές αρχές. Στον τομέα της, τραπεζικών η αξιολόγηση της ισοδυναμίας της χώρας περιορίζεται σε τρεις συγκεκριμένους ε, τομείς. Ε, πρώτα απ' όλα στο, στην στάθμιση, χαμηλότερη στάθμιση κινδύνων. Ε, οι διατάξεις ισοδυναμίας CRR δίνουν τη δυνατότητα στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουν αυτό το ζήτημα έτσι ώστε να είναι είναι καλύτερη η έκθεση, η κάλυψη μάλλον και μικρότερη η έκθεση σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Είτε πρόκειται ε, για φορείς όπως κεντρική τράπεζα, κεντρική ε, κυβέρνηση, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ. Το δεύτερο στοιχείο ε, είναι το απόρριτο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να καλούμε εποπτικές αρχές από τρίτες χώρες να συμμετάσχουν σε διαδικασίες επιτήρησης ή κολέγια επιτήρησης τα οποία έχουν οριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για διασυνοριακές, ας πούμε, για διασυνοριακούς τραπεζικούς ε, ομίλους κτλ. Αυτό μπορεί ε, να χρησιμοποιηθεί βεβαίω και να υλοποιηθεί πάντα μέσα σε όρους επαγγελματικού απορρίτου. Το τρίτο, η τρίτη το τρίτο στοιχείο αναφέρεται στην επιλογή που έχει η αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην χρησιμοποιήσει ε, ε, η ιδιαίτερη επιτήρηση consolidated supervision για τις ε, τραπεζικούς ομίλους τρίτων χωρών βάσει του άρθρου 127 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή όταν οι δομές είναι παρόμοιες. Η αξιολόγηση, οι αξιολογήσεις της ε, ισοδυναμίας γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μερικές φορές ε, ε, μετά και βάση και της πραγματογνωμοσύνης και της τεχνικής γνωμοδότησης και συμβουλής των υπηρεσιών των ευρωπαϊκών ε, εποπτικών αρχών. Με αυτή την έννοια τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 22 ε, έλεγχοι βάσει του CRD ε, και έχουν ελεγχθεί 34 αρχές. Ε, η, Κεντρική Τράπεζα κάνει, η, Τραπεζική Εποπτική Αρχή ε, συμμετέχει σε τέτοιες ε, αξιολογήσεις ισοδυναμίας χωρίς όμως να συμμετέχει σε όλη την διαδικασία. Εννοούμε ότι η επικοινωνία με τις χώρες, τις τρίτες χώρες αυτές σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί το, η απαραίτητη πληροφόρηση όσον αφορά το τεχνικό, ε, νομοθετικό ε, και λοιπό ε, πλαίσιο και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί μία χωρίς τέλος ισοδυναμία ή δυνατότητα χωρίς χρονικό περιορισμό δράσης στην ενιαία αγορά. Επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την δυνατότητα μετά από την ε, ε, έγκριση κάποιων τροποποιήσεων να αποσύρει ε, την ισοδυναμία. Παρατηρούμε ότι σε πολλές διασυνοριακές δραστηριότητες μπορεί να υπάρξουν ειδικέ συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό το έχουμε δει και σε πρόσφατα παραδείγματα όπως ας πούμε και στο πρόσφατο παράδειγμα ε, της, ε, του διαχωρισμού του CRD που μειώνει το πεδίο εφαρμογής ε, για την επιτήρηση όσον αφορά την φερεγγιότητα και επομένως δίνει την δυνατότητα σε τρίτες χώρες να έχουν την δυνατότητα πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ να ξεπεράσουν αυτού του είδους τους περιορισμούς. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει 30 δις συγγνώμη. Ε, ε, ε, πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να ανασκευαστεί η φερεγγιότητα καθώς επίσης και η ανθεκτικότητα όσον αφορά τα συστήματα ισοδυναμίας και επομένως να δοθούν κάποια διεθνή πρότυπα όσον αφορά την προληπτική εξέταση ισοδυναμίας. Επίσης θέλω να επαναλάβω ότι ο έλεγχος της ισοδυναμίας δεν γίνεται άπαξ και ισχύει για πάντα. Ε, πρόκειται για μια διαδικασία ε, η οποία ε, διαρκώς ανανεώνεται και διαρκώς αλλάζει και επομένως θα πρέπει και τα κράτη, οι τρίτες χώρες να συζητούν και με τις ε, ε, αρμόδιες ε, αρχές έτσι ώστε να κατανοούμε πλήρως την κατάσταση και να κατανοούμε κάθε φορά την αλλαγή των στοιχείων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Γκαμπριέλ Μπερναρντίνο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή σας που μας κάλεσε εδώ σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων για την ισοδυναμία. Αναγνωρίζοντα την ε, διεθνή φύση των ασφαλιών, η Κομισιόν αποφάσισε για την συνδυναμία τρίτων χωρών ε, για τα προληπτικά καθεστώτα και την φερεγγιότητα με την οδηγία φερεγγιότητα 2. Στόχος δεν είναι μόνο η επαρκής ε, προστασία και να μειωθούν τα αριθμιστικά κενά, αλλά να μην υπάρχουν και άλλοι επικαλύψεις. Ο ρόλος της ε, ΕΟΠΑ καθορίζεται στα ανάλογα άρθρα και στον κανονισμό της ε, ΕΟΠΑ. Στην ασφάλεια δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μία αξιολόγηση ισοδυναμίας. Η Οδηγία Φεργιότητας 2 προβλέπει ήδη τρεις, ε, τρία διαφορετικά είδη για την φερεγγιότητα του ομίλου και τον υπολογισμό της και την αντασφάλιση. Οι αποφάσεις αυτές ε, μπορούν να γίνουν για μια απεριόριστη περίοδο, για μια τρίτη χώρα αν θεωρηθεί πλήρως ε, ισοδύναμη, αλλά και για μια πιο περιορισμένη περίοδο. Βεβαίω, για να υπάρξει απόφαση πλήρου ισοδυναμία, θα πρέπει το καθεστώ τη ε, τρίτη χώρα να πληρεί κάποια κριτήρια, όπω αυτά αναφέρονται στην σχετική οδηγία και στα εφαρμοστικά μέτρα. Ο στόχο είναι να αξιολογήσουμε αν από την σκοπιά κάποιο ο οποίος έχει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, το αποτέλεσμα το οποίο επιτυγχάνεται είναι παρόμοιο με αυτό το οποίο επιτυγχάνεται με την Οδηγία Περιφερειακότητας 2. Τα κριτήρια βασίζονται στις γενικές αρχές του πλαισίου της δεύτερης οδηγίας και περιέχουν ζητήματα διοίκησης, ε, εποπτικών εξουσιών, διαχείρισης του κινδύνου, επαγγελματικού απορρίτου και βεβαίως τις ε, κεφαλαϊκές απαιτήσει. Οι αξιολογήσεις βασίζονται στο αποτέλεσμα και λαμβάνουν υπόψη την αρχή της ε, επικουρικότητας. Για να αξιολογήσουμε την ε, ισοδυναμία έχουμε σημαντικές απαφές με υποπτικές αρχές τρίτων χωρών και βεβαίως αυτή η συνεργασία έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να διατηρηθεί. Κυρίως οι αξιολογήσεις βασίζονται σε απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και σε όσα μας λένε οι υποπτικές αρχές τριτών χωρών, αλλά για την πλήρη ισοδυναμία επίσης η ΕΟΠΑ κάνει και επιτόπιες επισκέψεις στην τρίτη χώρα για να αντιληφθεί καλύτερα την εποπτική προσέγγιση και την εφαρμογή του κανονισμού. Η ισοδυναμία και οι αξιολογίες καθώς περιέχουν ποιοτικές κρίσεις απαιτούν πολλούς πόρους της ΕΟΠΑ και τις τρίτες χώρες. Παρ' θεωρούμε πως ε, η δουλειά που γίνεται έχει πάρα πολύ μεγάλο όφελος για μια κοινή αντίληψη διαφορετικών ρυθμιστικών καθεστώτων για να προωθήσει την σύγκληση και να υπάρχουν διεθνή τέτοια πρότυπα. Η ΕΟΠΑ έκανε τρεις πλήρεις αξιολογήσεις ισοδυναμίας ε, και κατόπιν ετήματος της Κομισιόν 12 αναλύσεις του κενού όπως ε, λέγεται σύμφωνα με την οδηγία Omnibus επιπλέον κάναμε άλλες 11 αξιολογήσεις ε, που εστίαζαν συγκεκριμένα στα, στο επαγγελματικό απόρριτο και τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω κάτι το πολύ σημαντικό της σημασία των τακτικών αξιολογήσεων. Υπάρχουν σαφείς ε, ρήτρες αναθεώρησης ε, και στην οδηγία και στις πράξεις κατεξιοδότησης στο μέλλον, σύμφωνα με το ότι η ΕΟΠΑ θα περάσει από την ρύθμιση στην εποπτεία. Έχει σημασία να παρακολουθούμε όχι μόνο τις ρυθμιστικές εξελίξεις σε τρίτες χώρες, αλλά και την πραγματική εφαρμογή των προσεγγίσεων αυτών. Για να κληρώσουμε τον ρόλο μας αυτό, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας η ΕΟΠΑ θα έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Και νομίζω αυτό θα παίξει μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να κάνουμε αυτές τις τεχνικές αναλύσεις και βεβαίως να παρακολουθούμε τα καθιστώτα τρίτων χωρών και ελπίζουμε ε, να ληφθεί υπόψη το ότι αυτό απαιτεί και πόρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Στίβεν Μαγιόρ. Τώρα έχει τον λόγο ο πρόεδρος της ΕΣΜΑ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής σας ε, που οργάνωσαν αυτήν την ακρόαση. Θα υπάρξουν κάποιες ε, επαναλήψεις και στα δικά μου σχόλια. Να ξεκινήσω. Γιατί είναι τόσο σημαντικό το θέμα της ισοδυναμίας. Πρώτα απ' όλα γιατί οι αγορές είναι παγκόσμιες, ε, αλλά τις εποπτεύουμε είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο και αυτό προφανώς εγείρει ζητήματα συντονισμού και Συνέπειε και γνωρίζουμε πω οι κίνδυνοι στι ε, χρηματαγορέ είναι διασυνοριακοί και μπορούν να ταξιδεύουν και πρέπει να συνεχίσουν να είναι σταθερές οι αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην επηρεάζονται αρνητικά από κινδύνους εκτός της Ένωση. Τώρα μάλιστα είναι κατάλληλη στιγμή να γίνει ένας απολογισμό ε, του συστήματο ισοδυναμία ε, του πώς αποδίδει, όπως αναφέρθηκε το τρέχον διεθνές περιβάλλον αλλάζει σημαντικά και επιπλέον έχουμε τώρα σημαντική εμπειρία με την εφαρμογή των συστημάτων ισοδυναμίας από όταν ε, είχαμε αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις μετά την οικονομική κρίση. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω το έγγραφο εργασίας της ε, Κομισιόν και να επισημάνω ότι δεν έχουμε ένα σύστημα ισοδυναμίας, έχουμε πολλά συστήματα ισοδυναμίας τα οποία όλα διαφέρουν ελαφρώς. Κάποια λέγονται ισοδυναμία, κάποια άλλα λέγονται έγκριση και υπάρχουν και κάποια άλλα που λέγονται στοιχεία ισοδυναμίας ή διαβατήρια τρίτων χωρών. Το κοινό στοιχείο λοιπόν σε όλα αυτά τα συστήματα είναι ότι μετά από μια αξιολόγηση βασιζόμαστε στις ρυθμιστικές αρχές της οικίας χώρας ε, και είναι βεβαίως μια αξιολόγηση που κρίνει το αποτέλεσμα. Δεν κοιτάμε γραμμή-γραμμή ταυτόσιμη νομοθεσία. Επίσης πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποια σημεία τη δικής μας νομοθεσία δεν έχουν ισοδυναμία, π.χ. αν δούμε τον τομέα των usage. Ε, όσον αφορά λοιπόν τον ρόλο της... Ε, όσον αφορά λοιπόν τον ρόλο των δικό μας, έχουμε κάνει κάποιες αξιολογήσεις, όπως ήδη αναφέρθηκε, από τον Ολιβιέ δίνουμε σύμβουλες ε, για τον Αμύρ, για τα Σιερά και όπως ε, είπε και η Κομισιόν ε, έχουμε τώρα 26 υπηρεσίες τρίτων χωρών και 20 αξιολόγησης που έχουν αναγνωριστεί από την ΕΣΜΑ και έχουμε πάνω από 30 μνημόνια συναντήληψης, πάνω από 1000 μνημόνια συναντήληψης που έχουν συνυπογραφεί με αρχές ε, άλλων χωρών, όπως ανέφερε και ο Ανδρέα, είναι ένα σύστημα το οποίο απαιτεί πόρους και χρόνο. Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος των συστημάτων ισοδυναμίας. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε μια συνεπή εποπτεία και ρύθμιση σε όλο τον πλανήτη. Δεύτερον, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ελέγχει τους κινδύνους που δημιουργούν όσοι συμμετέχουν στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες και τρίτον θα πρέπει να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο και να είμαστε μια ανοιχτή αγορά όπου και οι συμμετέχοντες εκτός της Ένωσης να μπορούν να συμμετέχουν. Σαφώς τα τρέχοντα συστήματα έχουν κάποια ωφέλη. Είμαι σίγουρο ότι τα τωρινά συστήματα ισοδυναμίας έχουν δώσει κίνητρα σε τρίτες χώρες για να συγκλίνουν προς τις δικές μας ρυθμιστικές απαιτήσεις και βεβαίως ε, μας βοηθά να αποφύγουμε επαναλήψεις ε, και ασυμφωνίες ε, γιατί βασίζεται στις ρυθμιστικές αρχές των τρίτων χωρών. Όμως είναι σαφές ότι θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό να δούμε πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα και να αντιμετωπίσουμε τυχόν ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα, υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία και βεβαίως οι αγορέ ε, διαφέρουν ε, όσον αφορά και τα επιχειρηματικά του μοντέλα, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι λογικά δεδομένων και των ε, διαφορών που υπάρχουν, αλλά παρόλα αυτά μια ευθυγράμμιση θα ήταν υποφελής. Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε ήδη στο έγγραφο εργασίας της Κομισιόν, μέχρι στιγμής γίνεται μια άπαξ αξιολόγηση και καλό θα ήταν να συνεχιστεί αυτή η παρακολούθηση ε, για το εάν πληρούνται τα καρτήρια ισοδυναμίας ε, και είναι πολύ θετική η πρόταση της Κομισιόν να εμπλέκονται οι αρχές ε, για την ένταση πόρων που απαιτούνται, αυτό αναφέρθηκε ήδη και θα πρέπει να πω για, τις, για τι οντότητε εκείνε που πρέπει να εγγραφούν στην Ένωση θα πρέπει να πληρώνουν ένα τέλο ε, στι ε, αρμόδιε ε, αρχέ, όπω πληρώνουν και όλε οι άλλε εποπτευόμενε οντότητε. για να καλυφθεί ένα μέρο του κόστου Να αναφερθώ σε άλλα δύο θεμελιώδη ζητήματα, τα οποία αναφέραμε ήδη στην έκθεση αναθεώρηση του ΕΜΗΡ του 2015. Πρώτα απ' όλα, γεγονό παραμένει ότι σε αυτή την φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει αυτό το σύστημα, ενώ οι άλλε δικαιοδοσίες τρίτων χωρών δεν το εφαρμόζουν. Και έτσι καταλήγουμε σε μια άνηση κατάσταση για οντότητες τη Ένωση σε σύγκριση με οντότητες τρίτων χωρών που ωφελούνται από το ότι δεν υφίστανται πολλά συστήματα εποπτικά ενώ συμμετέχουν στην ε, αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εγγραφούν και εκτός της Δεύτερον υπάρχει το ζήτημα το οποίο επίσης αφορά την αναλογικότητα και το μέγεθος ε, των ε, χρηματαγορών των τρίτων χωρών και της, ε, των κεφαλαίων αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, κατά πόσο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα ελέγξουν τους κινδύνους των συμμετεχόντων από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στην αγορά της Ένωσης. Στην πραγματικότητα βασιζόμαστε σε στις αρχές των τρίτων χωρών και οι ρυθμιστικέ αρχές της Ένωσης δεν έχουν τις δυνατότητες συλλογή πληροφοριών για να αξιολογήσουν αυτούς τους ε, κινδύνους και κατά κανόνα δεν έχουν τα εργαλεία που χρειαζόμαστε. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις των Ευρωβουλευτών για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Uh, Ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας πολύ ενδιαφέρουσες, πολύ χρήσιμες και προφανώς επιβεβαιώνουν την σημασία και την επιτυχία αυτού του καθεστώτος. Παράλληλα, υποδεικνύουν και διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν περισσότερο. Όχι μόνο ότι χρειαζόμαστε και πόρους αλλά και χρόνο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, αλλά και το τελευταίο σημείο που τόνισε ο συνάδελφος, ότι υπάρχει απουσία αμοιβαιότητας. και ότι οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές έχουν περιορισμένες δυνατότητες να αξιολογήσουν την επίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν οι φορείς αυτοί και αναγκαζόμαστε να βασιστούμε στις εποπτικές αρχές των τρίτων χωρών. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ξεκινάμε τώρα με τις ερωτήσεις. Για λόγους χρόνου πρέπει να ομαδοποιήσουμε τις παρεμβάσεις. Θα ξεκινήσουμε με τέσσερις ε, παρεμβάσεις. Ο κύριος Βάλς είναι ο πρώτος. Δύο λεφτά ο κάθε ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν άκουσα από κανέναν από τους ομιλητές μας οτιδήποτε για το Brexit και για το τι σημασία και πώς θα επηρεάσει την ε, ισοδυναμία. Μια ερώτηση λοιπόν γι' αυτό. Ξέρουμε ότι για πολλές από τις συναλλαγές ε, με διασυναριακό χαρακτήρα και αυτές που γίνονται σε ευρώ ε, ο συμψηφισμό γίνεται από γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε ανησυχίε για το μέλλον αυτών των ε, συναλλαγών αυτή τη στιγμή ε, προκύψει, γίνει το Brexit. Θα πρέπει να προσαρμοστεί η νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζει ότι η εποπτεία των συναλλαγών σε παράγωγα με, σε ευρώ ελέγχεται. Ένα σύστημα εποπτεία, ισοδυναμίας λένε ορισμένοι, θα ήταν μια εναλλακτική λύση. Τι λέει η Κομισιόν. Θα μας δώσει αρκετές εγγυήσεις στο σύστημα ισοδυναμίας, ούτω ώστε να έχουμε υψηλής ποιότητας μακροπροληπτική εποπτεία. Δεύτερη ερώτηση. Για κάποιους συμμετέχοντες στην αγορά, στον, δρόμο, στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το πρόβλημα είναι ότι με την ισοδύναμη η Κομισιόν μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αναστείλει το καθεστώ ισοδυναμία σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Ε, αυτή η ανησυχία είναι θεμητή και πώ μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα ισοδυναμία, ε, ούτω ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο Λιβιέ και ο Στίβεν νομίζω είναι οι αρμόδιοι για να απαντήσουν ε, σε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά μια και είπα τέσσερις θα συνεχίσω με την Περβάνς. Ε, και έτσι, αν συνεχίσετε όμως πρώτα θα, θα επιλέγουν στο τι θα απαντάνε. Να ξαναχρησιμοποιήσω τον όρο Brexit. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση χωρίς να σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που καθορίζεται από τον Brexit. Τρία σημεία θέλω να κάνω. Το θέμα της αναλογικότητας. Νομίζω ότι είναι ε, ένας όρος ανάλογος με την επικουρικότητα και τα λοιπά πασπαρτού ας πούμε χρησιμοποιήθηκε σε όλο το δυναμικό του και μήπως θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί, να επανεξεταστεί, να επανερμηνευτεί υπό το φως του Brexit. Δεύτερον, σε ορισμένε νομοθεσίες που, ή μάλλον νομοθετήματα ε, που είναι υπό εξέταση, θα τεθεί το θέμα της ισοδυναμίας. Το ισχύον σύστημα είναι περιπτωσιολογικό. Ε, όμως, δεν θα πρέπει να έχουμε δεν θα έπρεπε να έχουμε μία οριζόντια προσέγγιση για να επαληθεύσουμε το πώς ε, αντιμετωπίσουμε το θέμα των ισοδυναμιών, ειδικά με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ή, εν πάση στη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, το θέμα της ισοδυναμίας ισοδυναμιών θα τεθεί ως σημαντικό στοιχείο. Ε, πριν μπούμε στα επιμέρους νομοθετήματα, θα πρέπει να δούμε δηλαδή αυτό το στοιχείο της ισοδυναμίας με το Ηνωμένο ε, Βασίλειο. Στην ανακοίνωσή της η Κομισιόν ε, θέτει και το θέμα της απόσυρσης του, του καθεστώτος ισοδυναμίας. Πώς μπορεί να ξεκινήσει. Πώς ξεκινάει η διαδικασία. Φαντάζομαι... Να, ότι θα πρέπει να γίνει μια νέα εφαρμοστική πράξη. Ε, σωστό είναι αυτό. Δεν θα έπρεπε εν αυτή περιπτώσει ε, να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ξεκινήσει αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αντιπρόεδρος μας, η κυρία Σουίνμπορν. Μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, δεν θα σας εκπλήξει και τους εμπειρογνώμους δεν θα τους εκπλήξει. Και αφορά το, την πρόσφατη απόφαση ισοδυναμίας CCP μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, της, και των ΗΠΑ. Ο κύριος Μάγιορ και ο κύριος Γκόσαμ μπορεί να θέλουν να απαντήσουν. Στην περίπτωση της EFCSTC δεν έγινε μια απλή αξιολόγηση των κανόνων CFTC. Η Κομισιόν υπησύλθασε λεπτομέρειες ε, και αξιολόγησε ένα τελείως διαφορετικό σύστημα το δικό μας. Ε, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό νομικό πλαίσιο, για, μια, για ένα πλαίσιο αυτορύθμισης κτλ. Γενικά αναγνωρίζεται ότι υπήρχαν θέματα ανταγωνισμού ε, που ήταν τμήμα των διαφορετικών κανόνων. Και αυτό επηρέασε την τελική απόφαση της Επίση, υπάρχουν και διαφορέ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ότι είναι αυτή. Τα δύο καθεστώτα δεν μοιάζουν καταρχά. Ε, το θέμα τη ρευστότητα. Ε, και αν δεν ε, ε πάρουμε τη σωστή απόφαση, θα υπάρξει ε, ροή κεφαλαίων από το, τη χώρα ή από τη δικαιοδοσία με την υψηλότερη ροή κεφαλαίων προς αυτήν με τη μικρότερη. Επίσης, το θέμα της μόχλευσης δεν το αντιμετωπίσαμε σωστά. Θα πρέπει οι πιέσει ε, ανταγωνισμού από την αγορά να παίξουν οποιοδήποτε, οποιοδήποτε ρόλο στις διαπραγματεύσεις ισοδυναμίας ή θα πρέπει να βασιστούμε στα θέματα ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ε, συμπεριφοράς των αγορών. Επίσης, ε, επίσης μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με τη ρευστότητα. Ακούγοντάς σας, ε, θα πρέπει να μάθουμε τίποτα από αυτή την πιο ε, δημόσια απόφαση ισοδυναμίας μέχρι στιγμής και μήπως ε, το νομοθέτημα Omnibus θα μπορούσε ε, να βελτιώσει τις αποφάσεις δυναμίες, να τις κάνει λιγότερο κατακαιρματισμένες. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημα μου αφορά την ε, ε, ε επιτήρηση των CCPs. Πριν από λίγο καιρό η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή αποφάσισε ότι για λόγους ε, θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινό παρονομαστής. Αυτό όμως έχει, ε, θα έχει οπωσδήποτε επίπτωση ε, στα στοιχεία τα οποία βρίσκονται εκτός ε, ευρωζώνης ε, και ε, επομένως εγώ ρωτώ έχει αυτή η αρχή την ε, δικαιοδοσία για να παίρνει τέτοιες αποφάσεις και επίσης υπό τον κανονισμό EMI They have equivalent. Υπό τον κανονισμό ΕΜΙΡ ε, υπάρχει δυνατότητα ε, αναφοράς αυτών των στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως μετά τον Brexit ε, ενδεχομένως θα υπάρξει μια σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά τους ECPs εκτός Ευρωζώνης. Όμως συστηματικά σημαντικοί όγκοι θα εξακολουθούν να διακινούνται. θεωρούν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το συμπέρασμα ε, του 2011 είναι σωστό ή ε, ε, η κεντρική εποπτική αρχή έχει σκοπό να δώσει μεγαλύτερες δικαιοδοσίες στην Κεντρική Τράπεζα και γενικότερα τι πρόκειται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν μιλάμε για σημαντικές συστημικές αξίες. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα ερωτήματα, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Γκερσάν θα απαντήσει πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε όλη τη μέρα μπροστά σα και θα προσπαθήσω τουλάχιστον να ομαδοποιήσω κάποιες ερωτήσεις και ε, κάποιες απαντήσεις. Οι δύο πρώτοι ομιλητές ε, ε, αναφέρθηκαν ε, και οι δύο στην δυνατότητα του, της Ευρωζώνης να ξεπεράσει και να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Ε, κοιτάξτε, μάλλον πρώτο ετέθη το θέμα της δικαιοδοσίας της Κεντρικής Τράπεζας. έφυγε η, η κυρία η οποία έθεσε το ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει, ε, δεν θα το απαντήσω λοιπόν για να κερδίσουμε και χρόνο. Ε, και μετά είχαμε και την έρωση του κ. Μπόλτς. Κοιτάξτε, ναι, όντως ε, υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι σχεδίζεται ε, με τα Euro Denominated Instruments ε, και το κεντρικό θέμα με την Κεντρική Τράπεζα είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη δικιά της πολιτική και εγώ δεν μπορώ να κάνω κρίση πάνω σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει το άρθρο 22 του καταστατικού της Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να διαφωτίσει ε, επί του θέματος. Ε, αλλά ε, νομίζω ότι για την ώρα δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε με αυτό. Ξέρετε ότι βράχει πρόθεσμα η ομοφωνία είναι σημαντική. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να ξαναθέσω το ερώτημα αυτό με λίγο διαφορετικό τρόπο. Γιατί ξέρετε, στην ουσία αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ε, ποια είναι τα ποσά των συστημικών κινδύνων τα οποία επιτρέπεται σε κάποιον άλλον να ε, διαχειρίζεται. Ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να εμπιστευτούμε και τους ε, αντισυμβαλόμενους μας ε, και επομένως εάν εμείς πούμε δεν θέλουμε κανέναν ε, κίνδυνο και καμία διαχείριση κινδύνων στην ουσία θα αυξάναμε τον κατακαιρματισμό πράγμα κακό για την οικονομία έτσι κι αλλιώ. Όμως υπάρχουν όρια ε, σχετικά με το ε, τι μπορείς να επιτρέψεις ε, όσον αφορά διαχείριση κινδύνου εκτός των δικαιοδοσιών σου. Ε, και ε, πρέπει να ελέγξεις ποιους είσαι σε θέση και ποιους μπορείς να εμπιστευτείς. Ε, καταλαβαίνω ότι σημαντικό στοιχείο για τη συζήτηση είναι το θέμα των ΗΠΑ, αλλά ήταν σημαντικό και από τις δύο πλευρές. Κάποια πράγματα θα πρέπει να ξεκαθαριστούν όσον αφορά την δυνατότητα διαχείρισης κινδύνου και την διαλειτουργικότητα, γιατί ε, στο τέλος της ημέρας αυτό που ενδιαφέρει είναι οι πολιτικοί θεσμοί να έχουν την ε, δυνατότητα να δράσουν και σε αυτόν τον τομέα και επομένως αυτός είναι ένας κεντρικός στόχος. Αυτό που προσπαθούμε ε, να κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, εφαρμόζουμε τις αποφάσεις ισοδυναμίας και αυτό φαίνεται και στο έγγραφο εργασίας είναι ότι προσπαθούμε να έχουμε μία, μία διαβαθμισμένη προσέγγιση του θέματος έτσι ώστε να ξέρουμε ποια είναι τα τμήματα του κινδύνου τα οποία μπορεί να διαχειριστεί η τρίτη χώρα και ποιο, ποιος είναι ο βαθμός κινδύνου που μπορεί ε, βεβαίως φτάνει ένα επίπεδο, φτάνει ένα σημείο στο οποίο δεν μπορεί πλέον να γίνει αποδεκτός ο κίνδυνος. Τώρα το ποιο είναι αυτό το σημείο, ναι αυτό είναι συζήτηση και πολιτική. Αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα προφανώς. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένω να έχετε διαφορετική άποψη ή να έχετε ισχυρέ ε, απόψει όσον αυτό. Σε σχέση με την κυρία Μπερέσε Μα ακριβώς ε, για να μην είναι κενή νοήματος η αναλογικότητα ε, σαν έννοια προσπαθούμε να δουλέψουμε ε, με βάση την εφαρμογή της σωστής διαφάνειας έτσι ώστε ε, να έχουμε ένα τρόπο συνεκτικό και μη διακριτικό, δηλαδή που δεν οδηγεί σε διακρίσεις. Βεβαίως υπάρχει ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, αλλά αυτό το περιθώριο της διακριτικής ευχέρειας προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε ισοδύναμα. Αυτό ισχύει και για την απόσυρση. Ίσως να τα πω αγγλικά. γιατί όντως θα πρέπει να υπάρξει μια διασύνδεση και με τις εξουσίες που έχει η Κομισιόν όσον αφορά το θέμα αυτό. Εάν θέλει κανείς να είναι αξιόπιστος ε, στην διαχείριση των ισοδυναμιών, ιδιαίτερος δε λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο αυτή εφαρμόζεται, ε, γιατί ε, υπάρχουν κάποιες αλλαγές ας πούμε στις δικαιοδοσίες, στην νομική, ε, στην νομική ρύθμιση των ε, κρατών που τα βλέπεις απλώς να έρχονται και δεν έχεις δικαιοδοσία πάνω σε αυτά. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει οπωσδήποτε να, υπάρξει μια, ένας καλός βαθμός συνεργασίας με τις δικαιοδοσίες των άλλων χωρών. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε και σε θέση όμως να αντιδράσουμε γρήγορα σε οποιασδήποτε τέτοιες ε, αλλαγές. Και τότε ε, θα πρέπει να είμαστε σε θέση είτε να ε, αναιρέσουμε είτε να αποσύρουμε την ισοδυναμία. Ε, με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να υπάρξουν πολλές ε, συζητήσεις. Συμφωνώ βεβαίως ε, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή κατανόηση ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει και οπωσδήποτε η Κομισιόν με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσε να αποφασίσει μόνη της ή τέλος πάντων χωρίς να, χωρίς να δώσει την απαραίτητη πληροφόρηση να πάρει μια τέτοια απόφαση, να κάνει ένα τέτοιο βήμα. Αλλά Οπωσδήποτε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Το ίδιο ισχύει και ε, με, την, ε, ε, με την εγκατάσταση, με την, in, the true sense of it. με τη χορήγηση της ισοδυναμίας. με τον ίδιο τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί η διακριτική ευχέρεια και με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη συνένεση. Δεν απήντησα όλες Ερωτήσει ε, το ξέρω, αλλά βεβαίως μπορώ να επανέλθω εάν ε, υπάρξουν άλλες σχετικές ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Σχετικά με το CCPs και σχετικά με με το πώς διαφέρει η επιτήρηση όσον αφορά CCP τρίτων χωρών. Αυτό που είπε ο Ολιβιέ είναι σωστό. Δηλαδή υπάρχει υπό τον ε, ε, ισχύοντα μηχανισμό χορήγηση οδυναμιών η δυνατότητα να ληφθεί υπόψη η αγορά μιας ε, τρίτης χώρας. Ε, ε, σε αυτή την περίπτωση εμπίπτει και η εξέταση ισοδυναμίας των Ηνωμένων Πολιτειών ε, γιατί μπορεί να υπάρξουν στοιχεία τα οποία είναι διαφορετικά κυρίως όσον αφορά τα μέτρα για την σταθερότητα και είναι γεγονός ότι η ΕΣΜΑ έχει κάποιες επιπλέον εξουσίες αλλά χρησιμοποιεί τις εξουσίες αυτές μονάχα για τα αποκλίνοντα στοιχεία. Δεν έχουμε εξουσίες όσον αφορά ε, την αξιολόγηση των γενικών κινδύνων που ε, ε, μπορούν να δημιουργήσουν είτε στις επίσης των Ηνωμένων Πολιτών είτε άλλων τρίτων χωρών κινδύνους λέω μπορεί να δημιουργήσουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους νομοθέτες. Εμείς δεν έχουμε ιδιαίτερες εξουσίες, μπορούμε να ζητήσουμε πληροφορίες και κυρίως εστιάζουμε στην διαφοροποίηση βάσει των στοιχείων αυτών. Είναι νομίζω σημαντικό να δει κανείς ε, και τον τρόπο με τον οποίο άλλε δικαιοδοσίε ε, τη Ασία, α πούμε, ή εν προκειμένου ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, θα κινηθούν. Ζητούν, α πούμε, πλήρη καταχώρηση. Και οι συζητήσει των Ηνωμένων Πολιτειών πλήρω ελέγχονται από τους ε, ε, ε, Αμερικανούς νομοθέτες και επομένως πρέπει να, πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες αυτούς. Απλώς το σημείο κίνησης είναι διαφορετικό και πρέπει να πω ότι η ΕΣΜΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνει γνώση των περιθωριακών τροποποιήσεων ή αλλαγών και εν πάση περιπτώσει οι εξουσίες που έχει η ΕΣΜΑ όσον αφορά τα CCP ε, ε, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λίγο πιο περίπλοκες ας πούμε ή εξεζητημένες από ότι οι πληροφορίες που έχει για τα CCP τρίτων χωρών. Επίση. επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, όπως είπε και ο Λεβιό προηγουμένως, ε, είναι υπεύθυνη για την μικροεπιτήρηση και η, οποτεδήποτε οι απαιτήσει αλλάζουν, οπωσδήποτε λαμβάνονται υπόψη. Αυτή η διάταξη δεν υπάρχει στις ΗΠΑ, ούτε και στο Ηνωμένο Βασίλειο και γι' αυτό βλέπει κανείς και διαπιστώνει ότι τα μοντέλα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Από άποψη, ε, από άποψη μικροπροληπτικής ε, αντιμετώπισης ε, αυτή η Euroclearance μπορεί να είναι περιορισμένη γιατί βασίζεται μονάχα στις διαφορές και όπω η ερώτηση και ο Λιβιά αναρωτήθηκε προηγουμένως μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να ε, έχουμε γνώση όλων των αλλαγών που γίνονται σε μια άλλη χώρα και μέχρι ποιο βαθμό μπορούμε να τις ε, αξιολογήσουμε είναι διαφορετικό θέμα. Ε, όσον αφορά τα παράγωγα ιδιαίτερα, γνωρίζουμε και η Κομισιόν το ήξερε ότι, ε, ε, ότι εξαρτιόταν πολύ ο τρόπος με τον οποίο θα το αντιμεταπίζαμε και από τον τρόπο με τον οποίο ε, το θέμα αντιμετωπίζεται και σε επίπεδο ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρομαι των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως έπρεπε να το δούμε και από την ε, πλευρά της, και από τη σκοπιά της σταθερότητας. Όσον αφορά τώρα το κατά πόσον πρέπει να προχωρήσουμε προς νομοθεσία Omnibus, είναι λίγο δύσκολο το θέμα. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι θα πρέπει να δούμε ε, με προσοχή τον τρόπο με τον οποίο μπορούν ε, να βρεθούν ε, κοινοί παρανομαστές σε όλο το νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνοντα υπόψη ότι και η αντιμετώπιση και τα business models είναι διαφορετικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Περνάμε στην επόμενη. Στις επόμενες ερωτήσεις, Ματ Κάθι Δεν εδώ. Σβέν Γκίγκολτ. Σύντομα, Αυτό το οποίο πάντα με προβληματίζει και θα ήθελα να ακούσω και από εσάς ε, τις προσωπικές σας απόψεις είναι το εξής. Αν δούμε πόσο περίπλοκο ήταν να διασφαλίσουμε ένα παγκόσμιο επίπεδο εποπτείας ε, και ρύθμισης ε, στις 28 χώρες της Ένωσης και τώρα με τους κανόνες ισοδυναμίας ε, πάντα χρειάζεται καιρό για να ελέγξουμε την ομοθετική κατάσταση των εταίρων μας, ε, τις εποπτικές ε, πρακτικές τους και κάποια στιγμή χορηγείται ισοδυναμία. Πού βρίσκουμε τους πόρους να ελέγξουμε το πώς αλλάζουν τα παράγματα και πώς έχει πραγματική εφαρμογή. Πραγματικά αναρωτιέμαι πού βρίσκονται αυτοί οι πόροι. Πόσα άτομα έχετε για να κάνετε αυτή τη δουλειά. Η εντύπωσή μου είναι ότι δεν ε, καταφέρνουμε να έχουμε ούτε πραγματική εποπτική ρύθμιση ε, εκεί όπου έχουμε εποπτικές αρμοδιότητες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε πώς παρακολουθούμε όλες αυτές τις αποφάσεις, ε, τι πόρους έχετε. Δεν το έχω καταλάβει αυτό και φαίνεται πως είναι πλέον κρίσιμο το ζήτημα όσο πλησιάζουμε προς τον Brexit. Την στιγμή του Brexit προφανώς πριόρι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ισοδύναμο. Και μετά βεβαίω τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν σταδιακά και να απομακρυνθεί. Ε, πού είναι λοιπόν οι πόροι για κάτι τέτοιο. Θεωρείτε ότι έχετε τους ε, πόρους για να παρακολουθείτε τις ε, συστάσεις και αποφάσεις που λαμβάνετε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χάνεμανς δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μάτοκ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ στους ομιλητές. Να συγκρίνουμε την ισοδυναμία με τα παγκόσμια πρότυπα. Ορισμένε κριτικέ που ακούστηκαν για την ισοδυναμία είναι ότι το σύστημα είναι ευρωκεντρικό. Δηλαδή το στάτου ε, τη ε, ισοδυναμία το χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με απόφαση τη Κομισιόν και μπορεί να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή. Το είπε και ο κύριο Βάλ, ο συντονιστή μου στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα μπορούσαν να ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, να πιέσουμε να υιοθετηθούν παγκόσμια πρότυπα με ένα μηχανισμό απαραίτητο για να επιλύονται οι διαφορές. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ε, ολοκλήρωση των αγορών και τη δημιουργία μιας πραγματικά παγκόσμιας αγοράς. Ακούστηκαν πολλές κριτικές και εμείς κάναμε και είδαμε πολλές κριτικές. Παραδείγματο χάρη, το πλαίσιο τη Βασιλεία για τι τράπεζε είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού που λέμε. Η συγκεκριμένη μου ερώτηση λοιπόν είναι, θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα υιοθέτηση παγκόσμιων προτύπων ω εναλλακτική λύση στο στάτου τη ισοδυναμία σε ορισμένου άλλου τομεί ε, ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματο. Ευχαριστώ, Ιάκοπ Φον Βάιτσέκερ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που το παράδειγμα των ε, ΣΕΣΕΠΗ ήδη παίζει τόσο σημαντικό ρόλο των κεντρικών αντισυμβαλωμένων τόσο μεγάλο ρόλο στη συζήτηση και αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι ε, στο μέλλον μάλλον θα χρειαζόμαστε μια κλίμακα μεταξύ ενός εύρος του καθεστώτος ε, ισοδυναμίας τρίτης χώρας που θα πηγαίνει προς ε, την εξοεδαφικότητα και ως ε, τελευταίο ε, μέτρο τον επαναπατρισμό. Αν δούμε παραδείγματο χάρη τις προτάσεις περί διάσωσης και ανάκαμψης και την λυπή νομοθεσία, Ναι, βλέπουμε πως έχουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται με διακριτική ευχαίρεια και η... Και όπως είπε και ο Σβέν, δεν είμαστε τόσο προετοιμασμένοι και από πλευράς προσωπικού και για να διασφαλίσουμε ότι σε όλους τους σχετικούς ε, τομείς ε, θα έχουμε έναν ε, ενιαίο, μια ενιαία ευρωπαϊκή εποπτική αρχή, η οποία θα κάνει κουμάντο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα και εντό και εκτό κάποιοι να κάνουν αυτή τη δουλειά και να διαχειριστούν την διαδικασία. Πώ λοιπόν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, όπου οι ΙΠΑ ήδη χρησιμοποιούν την εξοδαφικότητα στο πλαίσιο τη τρέχουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο τη μεταρρύθμιση του ΕΜΗΡ για να έχουμε ένα παράδειγμα του πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα και ακριβώς να έχουμε αυτή την κλίμακα, όπως σας είπα, ένα φάσμα ολόκληρο. Ευχαριστώ τον Φαν Ντεκελάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία σύντομη ερώτηση για το μύθι και το ΜΥΦΙΡ. Θα πρέπει να έχουν υιοθετηθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 και βεβαίως γνωρίζουμε πως ε, αυτά αφορούν την εμπορία σε τρίτες χώρες και τις αποφάσεις ε, ισοδυναμίας. Το θέμα είναι αν εργάζεστε από αυτόν και πότε θα λάβετε αποφάσεις ε, ισοδυναμίας τρίτων χωρών για μύφιτ και μύφιτ. Σας ευχαριστώ. Ολυβιά Γκέρσα. Yeah, thank you. Um, the... <clears throat> On the question of... Ευχαριστώ για το θέμα των πόρων που έθεσε ο κύριος Γκίγκολτ. Αν θέλετε να σας πω ότι η DigiFisma θα πρέπει να έχει πάνω, πάνω από 308 θέσεις, ναι, εντάξει. Αυτό το οποίο προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι να περάσουμε από την νομοθεσία στην εφαρμογή και στην ε, κοινή αγορά, αλλά βεβαίως ε, και σε χώρες με τις οποίες εμπορευόμαστε. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό, γιατί θεωρούμε ότι ο κλάδος δεν θα επενδύει μακροπρόθεσμα αν υπάρχει αβεβαιότητα για τους κανόνες και θα πρέπει ακριβώ να δούμε το τι θα γίνει. Έχουμε ζητήσει στοιχεία με μια δημόσια πρόσκληση και δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ένα ένα, μια περιοχή αναθεωρήσεων όπου θα έχουμε συνεχώς ως 10, 7, 8, 9, 10 θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία και οι τρίτες χώρες με τις οποίες έχουμε κάνει συμφωνίες ε, ε, ισοδυναμίας. Έχουμε κρίνει ότι είναι ισοδύναμες. Θα είναι πράγματι ε, και θα παραμένουν ισοδύναμες. Βεβαίω αυτό αντλεί πόρους όχι μόνο δικούς μας αλλά και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών όταν μιλάμε για την εποπτική ισοδυναμία, νομίζουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. εντάξει, κάποια στιγμή. Βεβαίω, θα, ίσως θα πρέπει να επιλέξουμε. Εγώ θεωρώ ότι η ισοδυναμία είναι αναγκαία. Ε, αλλά βεβαίω ε, δεν ε, νομίζω ότι θα πρέπει να αποκοπούμε από τον υπόλοιπο κόσμο που παρέχει ρευστότητα στην Ευρώπη. Οπότε, εντάξει, ίσως κάποια στιγμή να μην υπάρχει επάρκεια πόρων, αλλά όχι τώρα. Το θέμα λοιπόν προσμήνων προδιαγραφών είναι ενδιαφέρον. Δεν είναι εναλλακτική είναι βάση. Εάν δεν έχουμε κάποιες παγκόσμιες προδιαγραφές δεν μπορούν να οριστούν ισοδυναμίες. Γιατί καταλήξαμε τελικά, όπως είπε, παρά το ότι βεβαίως όπως είπε και η κυρία το σύστημα διαφέρει σε πολλές πτυχές από τις ε, είπα. Μα γιατί έχουμε διεθνή ε, πρότυπα στα οποία έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, Αυτά είναι χρήσιμα για την ε, ισοδυναμία. Αλλά ε, τώρα είναι υποκατάστατο όχι. Και αν θέλετε να πιστείτε γι' αυτό. Αρκεί να σκεφτείτε μόνο το τίλακ. Ε, είναι τέσσερις σελίδες. Δεν ξέρω αν έχετε δει τελευταίω τις νομοθετικέ προτάσεις επί του ΤΙΛΑΚ. Είναι 60 με 70 σελίδες. Δεν είναι ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικό τόσο αποτελεσματική όσο συνάδελφοι στην FSB, αλλά πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές όταν νομοθετούμε που δεν ε, αναφέρονται ρητό σε διεθνή πρότυπα από την φύση τους. Οπότε δεν είναι υποκατάστατο. Και καμιά φορά ίσως ε, πάμε παραπέρα και αναρωτιέται κανείς αν δούμε την περίπτωση των IFRS ότι εμείς είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που έχουμε χωρίσει την κυριαρχία μας σε έναν διεθνή φορέα και είμαστε από τις λίγες ε, μεγάλες δικαιοδοσίες που εφαρμόζουν πλήρως τα IFRS. Τώρα αν είναι σωστό ή όχι δεν ξέρω. Για τις ε, ερωτήσεις του κυρίου Φων Βάιστσέκερ για το MIFID MIFIR. Ναι, το ε, εξετάζουμε, έχουμε στείλει ερωτηματολόγια σε χώρες που δείχνουν ότι έχουμε ενδιαφέρον. Βεβαίω ε, υπάρχει ενδιαφέρον για τον κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ισοδυναμία, μη και η τεχνική δουλειά συνεχίζεται. Οπότε προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι την 1η Ιανουαρίου 2018. Οπότε το η ερώτηση του κυρίου Φωνοβάης Τσέκερ. Όπως είπα, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αντικατοπτρίζεται καλύτερα στην υφιστάμενη νομοθεσία. Οι αρχές ε, που νομίζαμε ότι υπήρχαν εκεί αλλά έχουν αναπτυχθεί μέσω της ε, πρακτικής ε, των 220 των αποφάσεων. Τώρα, το αν υπάρχει ανάγκη μια γενικότερη αναθεώρησης, όπως είπε η κυρία Μπερές, μίλησε για ένα όμνιμπους, εντάξει, είναι δυνατόν, είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθούσε, δεν ξέρω. Ε, Υπάρχουν ε, πολλές επιλογές μεταξύ του τι κάνουμε, δηλαδή λέμε στον κόσμο ότι εμείς έτσι ερμηνεύουμε τις ε, διατάξεις ε, και έτσι τις εφαρμόζουμε και θεωρούμε ότι για την ώρα είναι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να υπάρξει κάποια ισοδυναμία. Τώρα βεβαίως υπάρχει περιθώριο συζητήσεων και στο μέλλον. Αν υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα τώρα το να μπουν όλα αυτά σε ένα κείμενο, αυτό κατά την απόψή μου είναι θέμα πολιτικής ε, κρίσης. η επιλογή μεταξύ του να είναι κανείς γρήγορος και αποτελεσματικός ή να είναι ε, όμορφος και οργανωμένος. Σας ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, από τις ε, τρεις εποπτικέ αρχές ποιο ε, θέλει τον λόγο. Γκαμπριέλ Μπερναρντίνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το θέμα που είπε ο κύριος Γκίγκολτ για την εποπτική σύγκληση και το θέμα των πόρων μας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα, προσπάθησα να το κάλυψω στην παρουσίασή μου. Ε, είμαστε σε μια κατάλληλη στιγμή και γι' αυτό υπάρχει αναθεώρηση του συστήματος EFSS ε, στην Ευρώπη έχουμε δυνατότητα να χτίσουμε πιο καλούς θεσμούς, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε την εποπτική σύγκληση. Το θέμα δεν είναι μόνο το θέμα της ισοδυναμίας με τρίτες χώρες, αλλά και της ε, εποπτική σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει προφανώς να έχουμε περισσότερους πόρους, ε, και να δώσουμε σε αυτό το τομέα τη εποπτική σύγκληση περισσότερους πόρου. Για το θέμα της ισοδυναμίας θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση αναλογικότητας και να κάνουμε ιεράρχηση. Δηλαδή στην περίπτωσή μας θα πρέπει να εστιάσουμε ε, στις περιπτώσεις που δίνουμε πλήρη ισοδυναμία. Γιατί στην πραγματικότητα τι κάνουμε. Λέμε στι υποπτικές αρχέ τη τρίτη χώρα, αυτέ είναι οι βάσει αξιολόγηση του κινδύνου ε, οι ίδιες δηλαδή με αυτές που έχουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε τους πόρους για να τους παρακολουθούμε και από εποπτική σκοπιά να βλέπουμε κατά πόσον εφαρμόζεται και πώς εφαρμόζεται αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός. Το θέμα δεν είναι μόνο το θέμα κανόνων, το θέμα είναι το πώς τους εφαρμόζεις και πόσο αποτελεσματικός είσαι, ε, το πόσο εξετάζεις σωστά τους κινδύνους και τη διαχείρισή τους για το κατά πόσο πρέπει να έχουμε παγκόσμια πρότυπα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Λιβιέ. Τα παγκόσμια πρότυπα δεν υποκαθιστούν τη διαδικασία της ισοδυναμίας. Ούτω ή άλλω υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία σε διαφορετικά θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στι ασφαλίσει, η παλιά διαδικασία ισοδυναμία που ξεκίνησε πριν από ε, μερικά χρόνια με κάποιε τρίτε χώρε, επειδή δεν υπήρχαν ε, ισχυρά παγκόσμια πρότυπα, για τις ασφαλίσεις, ε, η διαδικασία της ισοδυναμίας ήταν καταλήτης για να κλείσουν και κάποια παραθυράκια ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή αρχίσανε και τρίτες χώρες να, ε, να υφετούν αρχές που βρίσκονται στο Solvency 2, στην Φερεγγιότητα 2. Και τελικά βελτιώνονται κάπως τα πράγματα σύν το χρονού ώστε να φτιάξουμε υγιή και ασφαλή παγκόσμια πρότυπα. Οι ασφαλίσεις βέβαια λειτουργούν λιγάκι διαφορετικά γιατί δεν έχουμε παγκόσμια πρότυπα, αλλά όμως ε, η διαδικασία της ισοδυναμίας και εκεί αποδείχθηκε πολύ σημαντική διαδικασία. Ο Στίβεν. Να απαντήσω στα τρία θέματα. Καταρχάς, ε, το θέμα των πόρων. Το να ρωτάτε την, ε, τον πρόεδρο των ε, ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών αν έχουν ε, αρκετούς πόρους, τι να σας πω. Προφανώς χρειαζόμαστε αρκετούς πόρους ανάλογα ε, με το αν ελέγχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ή σε περιφερειακό επίπεδο κάποια πράγματα. Φυσικά θα πρέπει να δώσουμε πόρους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απαραίτητος πόρους για να γίνει αυτή η προσπάθεια. Για το θέμα της κλίμακας ε, που ανέφερε ο Τζέικο Βάιτσέκερ, από την πλήρη ισοδυναμία πάνω-πάνω μέχρι τον ε, επαναπατρισμό των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων κάτω-κάτω στην κλίμακα. Υπάρχουν και ενδιάμεσες λύσεις, μην ξεχνάμε. Έτσι. Πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουν ε, οι αρχές στις τρίτες χώρες όπου λένε μπορεί να κάνετε, ας πούμε, συμψηφισμό δολαρίων σε ευρώ, αλλά χρειαζόμαστε καταχώρηση και εποπτεία με, τους δικούς μας, με τις δικές μας εποπτικές αρχές. Θα πρέπει να δούμε τη δυνατότητα να έχουμε περαιτέρω εποπτικά μέτρα. Επιπλέον, το σύστημα ισοδυναμίας από μόνο του έχει πολύ σημαντικά ωφέλη, γιατί ενθαρρύνει και δίνει κίνητρα στις ε, τρίτες δικαιοδοσίες για να συγκλίνουν με τα δικά μας πρότυπα. Και σε μέρε περιπτώσεις θέλουμε να βασιζόμαστε 100% ε, στα συστήματα των τρίτων ε, δικαιοδοσιών γιατί είναι μικρότερες δικαιοδοσίες, μικρότερα εδάφη χώρε ή έχουν λιγότερη σημασία. Επομένως εγώ θεωρώ ότι έχει νόημα να προσπαθήσουμε σε κάποιο βαθμό να βάλουμε κάποια στοιχεία αυτού του, του συστήματος, του ξένου και να τα ενσωματώσουμε στο δικό μας. Για τη Άκουσα τα θετικά που είπε ο Λιβιέ για το θέμα αυτό και είναι σημαντικό να επιληθεί το θέμα αυτό πριν ξεκινήσει το 2018, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξωτερικό ε, θα πρέπει να είναι και το εξωτερικό έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είμαστε όλοι έτοιμοι ε, για την έναρξη του MIFID MIFIR αρχές του 2018. Προηγουμένως ε, καλά το είπε ο κύριος Φεν Κίγκολτ ε, ότι θα είναι ε, δύσκολη δουλειά της αξιολόγησης και δύσκολη εξισορρόπηση. Εν πάση περιπτώσει όσον αφορά την προληπτική ε, εποπτεία των ε, Ιδρυμάτων. Πρέπει κανείς να καταλάβει ότι η εποπτεία ε, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις δικές μας αρχές. Τα κύρια στοιχεία εδώ θα είναι τα εξής. Να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίες χορηγήσεων είναι σωστές, ότι υπάρχει αρκετή μόχλευση όσον αφορά ε, την παροχή υπηρεσιών όσον αφορά, ε, πληροφοριών για τις δραστηριότητες ε, της εταιρεία και ότι έχει γίνει σωστή αξιολόγηση κινδύνου. Όσον αφορά τώρα την Consolidated Supervision, υπάρχει η πρόταση της Κομισιόν έτσι όπως αναφέρεται στην αναθεώρηση του CRB και ε, ε, εκεί ε, αναφέρεται η δυνατότητα consolidated supervision σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως συχνά παραμελούμε το ζήτημα της επίλυσης και της δυνατότητας επίλυσης. Ας πούμε, σε περίπτωση κρίσης θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι σαφής η κατανόηση των κανόνων μας και είναι σαφής η αρμοδιότητα ε, των ε, δικαιοδοσιών. Νομίζω ότι και εδώ όμως ε, κάνουμε πολλές πρόοδους όσον αφορά τον σχεδιασμό επίλυσης και όσον αφορά ε, και την ε, ε, βαθμιαία αντιμετώπιση των διαφορετικών τρόπων επίλυσης. Βεβαίως κατανοούμε ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής της Βασιλείας μπορεί να είναι ιδιαίτερα υποβοηθητική γιατί ακριβώς βασίζεται στη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα. Ας πούμε σήμερα ο υπεύθυνο μας βρίσκεται στην Κίνα κάνοντας ε, την αξιολόγηση ε, για την ε, χώρα αυτή όσον αφορά συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επομένως, οπωσδήποτε λαμβάνουμε υπόψη διεθνή πρότυπα για την αξιολόγηση και της επίπτωσης που μπορεί να έχει η δικαιοδοσία και η νομοθεσία άλλων χωρών. Πολύ ωραία. Τελευταίος γύρος ομιλητών είναι η Ναγκίλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους για τις παρουσίασεις σας. Ε, ναι, το θέμα του Brexit. Given that there are... Το θέμα του Brexit ε, είναι κακιά λέξη, δεν την λέμε εύκολα, εν πάση περιπτώσει. Ε, νομίζω ότι πέρα από τις σημερινέ διαβουλεύσεις είμαι βεβαία ότι θα υπάρξουν, θα προκύψουν κάποιες νέες τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις. Αυτό που είναι σημαντικό, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση και αν ε, υπάρξει, ε, το σημαντικό είναι να μπορεί να λειτουργήσει και οπωσδήποτε θα πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία κάποιες υπεραπαιτήσεις. Ε, τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες υλοποιούνται πλήρως στις 27 ή 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει λόγος να φτάσουμε σε υπερβολές αυτό για το οποίο δεν είμαι σίγουρη είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε σε μια καλή ισορροπία, δηλαδή πώς μπορούμε να αποφύγουμε ιδιαίτερο βάρος για την επίτευξη της ε, ε, ε, μιας σωστής ισορροπίας. Επίσης, το θέμα των ισοτιμιών μπορεί να είναι και πολιτικό, δηλαδή πώς μπορεί η Κομισιόν να αποφύγει οποιαδήποτε πολιτικοποίηση εντό εισαγωγικών της χορήγησης ε, ε, ισοδυναμίας. Ε, επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και πιο αναλυτική η πρόσβαση στα δεδομένα και τα στοιχεία των τρίτων χωρών οπωσδήποτε. Αλλά αυτό μπορεί να περιέχει και ένα στοιχείο υποκειμενισμού και από την άλλη πλευρά χρειάζονται ιδιαίτεροι πόροι. Πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό και λαμβάνοντας υπόψη Ε, λαμβάνοντας υπόψη και το θέμα της, ε, ε, της, των, της, του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε πάνω από 300.000 προϊόντα, τα οποία προέρχονται από 5.000 περίπου και πλέον εταιρείε. Πώς είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλα αυτά. Ίσως θα πρέπει να βρεθούν κάποιοι άλλοι μηχανισμοί όσον αφορά την επιτήρηση των ε, CCP, ε, των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Ε, είναι κατανοώ τη θέση σας, όμως υπάρχουν και κάποιοι, κάποιες άλλες φωνές που λένε ότι ενδεχομένως θα υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά την ενωσιακή οικονομία και σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί η επιτήρηση. Thank you. Κύριο Στόλογεν. Ε, ευχαριστώ. Έχω μια απλή ερώτηση. Ε, υποθέσουμε ότι πλήρωνται όλα τα κριτήρια ισοδυναμίας από τον τραπεζικό τομέα σε μια χώρα, ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από δύο χρόνια. Μπορούμε τότε να αντιληφθούμε ότι η κατάσταση αυτή θα είναι παρόμοια με το να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο. Σημειώσατε ότι η Νίνα Τζίλ χρησιμοποίησε περισσότερο χρόνο, οπότε εσείς χρησιμοποίησατε λιγότερο. Τέλος, Πέντρο. Σίλβα Πέντρο. Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, ακούστηκαν πολλά πράγματα για την ισοδυναμία τρίτων χωρών και οι περισσότεροι συνάδελφοι βεβαίως ε, εξέφρασαν διάφορες ανησυχίες. Εγώ θα ήθελα να φέρω ένα ε, ζήτημα το οποίο αφορά το σύστημα της διάσωσης τραπεζών. Και εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια ανισότητα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια συνεπή αντιμετώπιση. Γνωρίζουμε πως η οδηγία για τη διάσωση των τραπεζών ε, δεν προβλέπει κάποια ρήτρα ισοδυναμίας, αλλά γεγονός είναι πως κάτι τέτοιο μπορεί να έχει διασυνοριακές επιπτώσεις και επιπτώσεις σε τρίτες χώρες, κυρίως όταν μιλάμε για τραπεζικούς ομίλους που δραστηριοποιείται παγκοσμίω. Αυτός είναι ο λόγος επίσης για τον οποίο θεωρώ πως υπάρχουν προβλήματα ισοδυναμίας τα οποία δεν έχουμε αντιμετωπίσει επαρκώς π.χ. η χρήση των ε, ενιών ε, των, των ε, φορέων εξυγίανσης ή των ε, άλλων ε, δομών που συνδέονται mm-hmm. ε, με αυτούς. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ξεκάθαρη μεταχείριση για τις υποεξηγένσεις τράπεζες και σε τρίτες χώρες και να δούμε σε ποιο βαθμό θα ήταν χρήσιμο να έχουμε κανόνες ισοδυναμίας και για αυτές τις περιπτώσεις. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορά το άρθρο 5 της οδηγίας ε, έχω τις επιφυλάξεις μου για το waiver αυτό για το bail-in και εδώ πέρα νομίζω τίθεται το ερώτημα μήπως στην περίπτωση μιας αμοιβαίας αναγνώρισης ή ενός συστήματος ε, ισοδυναμίας ε, θα μπορούσε να ε, χρησιμεύει κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα για το συνολικό πλαίσιο που έθεσε η υπερβάνωση Μπέρες. Μήπως χρειαζόμαστε ένα οριζόντιο σύστημα ισοδυναμίας. Και τελευταίο γύρος απαντήσεων ξεκινάμε με τον Ολιβιέ. Να έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Η πρώτη και η δεύτερη ερώτηση είναι ουσιαστικά ίδιες. Πρέπει να επαναλάβω κάτι που είπα στις αρχικές μου παρατηρήσεις. Η ισοδυναμία δεν σημαίνει ότι έχουμε τους ίδιους κανόνες κτλ. Η ισοδυναμία σημαίνει ότι, όπως είπε και ο κύριος Λατινσίλη είναι ένα φάσμα ολόκληρο εξαρτάται από το επίπεδο διασύνδεσης ε, που έχουμε και τη δυνατότητα και το, την πιθανότητα εισαγωγής κινδύνων από άλλες ε, χώρες και αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες μας δίνουν ε, τα ίδια αποτελέσματα όπως οι δικοί μας κανόνες και όσο βεβαίως ε, μεγαλύτερη διασύνδεση τόσο υψηλότερη κίνδυνη και όταν η διασύνδεση είναι πλήρης ε, πρέπει να είμαστε πολύ έχουμε μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνη συμφωνώ με την κυρία Γκίλ ότι ε, την πρώτη μέρα του Brexit οι κανόνες θα είναι οι ίδιοι και οι πρακτικές επίσης και βεβαίως Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κρυθεί μετά από πολύ προσεκτική ανάλυση. Αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορώ να πω. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν θα έχουν διαβατήριο οι Βρετανικές τράπεζες. Όχι, γιατί διαβατήριο πέρα από το IFMD, εκτός αν είναι ένα γλωσσικό ζήτημα, το διαβατήριο έχει κανείς όταν είναι εντός της ε, ενιαίας αγοράς και το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να μην είναι στην ενιαία αγορά. θα έχουν τη δυνατότητα ισοδυναμία σε βρετανικές τράπεζες. Θα δούμε, δεν έχω κάποιο λόγο να αμφιβάλλω. Ε, ο Ανδρέα υπενθύμησε τους τομείς στους οποίους υπάρχει ισοδυναμία. Και τέλος, αυτό το, αυτή την έννοια της Ευρώπης Φρουρίου δεν την αντιλαμβάνουμε. Γιατί εκεί που δεν υπάρχει ισοδυναμία είναι γιατί δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει η, η συμμεταχείριση με αυτούς που είναι στην ε, εσωτερική αγορά. Γιατί δηλαδή δεν χρειάζεται να δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτή η έννοια της Ευρωσουλίου δεν είναι κάτι που αντιλαμβάνομαι γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είμαστε πιθανότατα ε, η πιο ανοιχτή περιοχή του πλανήτη στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ε, θέσατε επίσης ε, το δάκλοπι των τύπων των ήλων ε, ότι πράγματι όταν κάτι δεν είναι μέρος της δικής μας της δικαιοδοσίας θα πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός εμπιστοσύνης ο οποίος θα είναι πολύ υψηλός ειδικά αυτά τα οποία είπαμε εμείς ε, για τις επιτόπιες επισκέψεις ε, κτλ. Ναι, ισχύουν αυτά και για τις ΙΠΑ ε, ναι, αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται πόροι και αυτό δείχνει ότι βεβαίως η νομοθεσία δεν είναι το μόνο θέμα που διακυβεύεται εδώ. Τότε όσο περισσότερο θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το μοντέλο σε σε χώρε με τι οποίε υπάρχει μεγάλος βαθμός ε, αλληλεπίδρασης νομίζω ε, τόσο περισσότερο θα απασχολήσει αυτό τι ευρωπαϊκέ αποπτικές αρχές, είναι σαφές. Ε, η τελευταία ερώτηση κυρίου Σίλβα Περέρα. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σύστημα εξυγένση τραπεζών, ισοδυναμία, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε σε περίπτωση εξυγένση είναι η συνεργασία, όχι η ισοδυναμία. Αν χρειαστεί ποτέ να εξηγιάνουμε έναν μεγάλο διεθνή τραπεζικό όμιλο, ε, δεν ενδιαφέρει. Τη είπα αν ε, θα είμαστε ισοδύναμοι και, ε, και, και εμά δεν μα ενδιαφέρει, να πω την αλήθεια. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί. Γιατί αν δεν καταφέρουμε να το επιλύσουμε από κοινού, τότε θα είναι ε, άσχημε συνέπειε για όλου. Γι' αυτό κάνουμε δοκιμέ με τις αρχές των ΙΠΑ και τα λοιπά. Δεν προβλέπουμε λοιπόν ένα σύστημα ισοδυναμίας γιατί πραγματικά δεν ελαμβανόμουν ποιος, ε, ποιον θα αφορούσε. Το θέμα είναι να εφαρμόζουμε τις διεθνείς προδιαγραφές ε, με τρόπο ενιαίο, ποιος θα κάνει τι σε περίπτωση προβλήματος και γι' αυτό έχουμε ακριβώς ε, τακτικές σκήσεις που κάνουμε ναι. με τους ε, συναδέλφους μας, ε, δεν τις δημοσιοποιούμε. Ε, εάν, ξέρω εγώ, η τράπεζα αντιμετωπίζει προβλήματα, γιατί θα κάναμε. Και δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Για το Μπέιλιν, το συμβατικό, δεν είναι πανάκια. Και πάλι η ισοδυναμία δεν θα βοηθούσε, νομίζω στόχο έχει να διασφαλίσουμε ότι ομόλογα σε ε, τρίτες χώρες ε, θα υποστούν και αυτά το Μπέιλιν. Και τελικά βεβαίως ε, υπάρχει και το θέμα της εκδοτικής ευχαίριας της κρίσης της εποπτικής αρχής. Και αν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ενιαίο Εποπτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι οι διαβεβαιώσεις αυτές δεν υπαρκούν, θα ζητούσε από τις ε, τράπεζες ε, να εκδώσουν ε, και κάποιες άλλες εγγυήσεις εάν θεωρούν ότι οι εξτάμενες δεν μπορούν να υποστούν bail-in. Νομίζω ότι δεν τίθεται ζήτημα ισοδυναμίας όπως αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Στίβεν Μαγιόρ και μετά Ανδρέα. Να αντιδράσω. Στο πρώτο σημείο που ακούστηκε, στο, επιχείρημα ότι η Ευρώπη είναι ένα φρούριο και ότι είναι δύσκολο να μπει κανείς στην Ευρώπη. Συμφωνώ με αυτά που πολύ Λιβιέ. Και να πω και κάτι που είπα και στην αρχική μου παρουσίαση. Τώρα είμαστε σε μια φάση όπου οι συμμετέχοντες στην ευρωπαϊκή αγορά, αν θέλουν να κάνουν ε, συναλλαγέ και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υποστούν πλήρη καταχώρηση. Μερικές φορές υπάρχει το υποκατάστατο της συμμόρφωσης, αλλά συνήθως υπάρχει πλήρης καταχώρηση, πλήρης εποπτεία. Εκτός, έτσι. Ενώ εμείς βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στις ξένε ξένες ρυθμιστικές αρχές. Η απόφαση ισοδυναμίας είναι σοβαρή απόφαση και αυτή τη στιγμή δοθεί η ισοδυναμία ε, είναι ένα μεγάλο βραβείο που παίρνει κανείς. Έχει ελεύθερη πρόσβαση, περιορισμένες, ε, περιορισμένο ε, ρυθμιστικό και εποπτικό κόστος κτλ. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι σωστό να λέμε ότι η Ευρώπη είναι φρούριο. Για το δεύτερο σχόλιο. Εμείς θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πιθανότητες για να αυξήσουμε τις εξουσίες που έχουμε, ώστε να παίρνουμε πληροφορίες από τις τρίτες χώρες και να έχουμε ε, και να, να βλέπουμε τι εποπτικά εργαλεία υπάρχουν στις ξένες εποπτικές αρχές για να ελέγχουν τους φορείς ε, που λειτουργούν εκεί. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τα ίδια που κάνουν και οι ξένες εποπτικές αρχές. Θα πρέπει να βασιστούμε και να ε, ελέγξουμε τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν εμάς. Το θέμα είναι, έχουμε παρκείς εγγυήσεις ότι οι ξένες εθνιστικές αρχές δίνουν την ίδια προτεραιότητα με τους κινδύνους που αφορούν εμάς ε, και επιπλέον, μην ξεχνάμε ότι έχουμε λίγους πόρους ε, και λογικό είναι οι εποπτικές αρχές, οι ρυθμιστικές αρχές μάλλον να εστιάσουν καταρχάς στους κινδύνους που αφορούν τη συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Ίσως υπάρχει και νομική υποχρέωση. Ε, είναι λογικό. Όχι... Επομένω, εμεί δεν θέλουμε να ξανακάνουμε τη δουλειά. θα βασιστούμε σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς αλλά θέλουμε να λάβουμε υπόψη μα στου κινδύνου που προκαλούν αυτοί, αυτές οι οντότητες όταν συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα, πώς ε, χρηματοδοτούμε. Ε, με τέλη. Ε, ε Παραδείγματος χάρη, ε, η οίκη αξιολόγησης, ας πούμε, ε, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την έγκριση δωρεάν. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Ε, θα πρέπει να ψάξουμε ε, να βρούμε ένα σύστημα που να βασίζεται στα τέλη. Όταν κάποιο έχει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, να απαιτούμε να καταβάλει κάποια τέλη. Ευχαριστώ. Ο Ανδρέα, να ενισχύσω αυτό που είπε ο Λιβιέ για το θέμα της εξυγίασης. Κατά τύχη, ε, είχαμε μια καλή περίπτωση, επιτεχή περίπτωση διαμεσολάβησης είχαμε ένα διασυνοριακό ε, σχέδιο εξυγίανσης και μάλιστα συμμετείχε και τρίτη χώρα. Σε αυτό το σχέδιο εξυγίασης, η συνεργασία και οι δομές που εξασφάλισαν ότι θα μπορέσεις να κάνεις, ε, να κάνεις το bail-in που απαιτείται και ότι υπάρχουν ε, και οι δομές, ούτως ώστε στην τρίτη χώρα να υπάρχει σωστή εξυγίανση, χωρίς προβλήματα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βεβαίως το, πόσο διασυνοριακό, το διασυνοριακότητα του ομίλου και να δούμε κατά πόσον έχουμε όμοια εργαλεία εμείς ε, και εκτός. Ε, όσο πιο όμοια είναι αυτά τα εργαλεία, τόσο πιο εύκολο είναι να βασιστούμε στο τι κάνουν οι αρχές στις τρίτες χώρες. Το βασικό είναι ότι ε, στα πλαίσια της BRD, ε, η BRD συγγνώμη, πρέπει έχουμε όλα τα εργαλεία, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις ε, των φορέων που δραστηριοποιούνται εντό της αγοράς μας. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ευχαριστούμε και την Κομισιόν και τους τρεις εκπροσώπους των φορέων Ήταν πάρα πολύ καλή και καρποφορά η συζήτηση. Υπό τα διάφορα δεν έχω κάτι. Δεν ξέρω αν έχετε εσεί κάτι να πείτε, όχι επόμενη συνεδρίαση την επόμενη Δευτέρα στις 8 το βράδυ ε, στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος της συνεδρίας.